Der Präsident! Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να με ακούσετε λιγάκι προσεκτικά. Θα λάβω ένα μέτρο που δεν το συνηθίζω να το κάνω, το θεωρώ όμως απαρέγκλητο για την τάξη που πρέπει να επικρατήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα το πρωί υπήρξε ένα επεισόδιο για το οποίο πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραμείνει άπραγο. Είναι υποχρεωμένο να αντιδράσει. Θα σας παραθέσω αυτό λεξί μία πρόταση που τη θεωρώ απαράδεκτη και που πρέπει να την τιμωρήσουμε. Παραθέτω αυτά που είπε ο συνάρφος κύριος Συναδεινός, ο οποίος ε, σήμερα το πρωί στη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είπε τα εξής και παραθέτω. Όπως έχουν γράψει Οθωμανοί επιστήμονες, οι ε, Τούρκοι είναι βάρβαροι, είναι βρώμικοι, οι Τούρκοι είναι όπως τα σκυλιά οι οποία γαβγίζουν, τα οποία γαβγίζουν και κάνουν τα ανίκητα, ε, όμως όταν έρθει ο εχθρός υποχωρούν. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι Τούρκοι μόνο με την πυγμή και την αποφασιστικότητα. Ε, τέλος της παράτασης. Άρα δηλαδή ε, πρόκειται κυρίες και κύριοι με βάση το άρθρο 165 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα οποία είναι προσιλωμένη και υποκλίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. κατόπιν τούτου ως ε, μέσο και μέτρο με συγχωρείτε το οποίο λαμβάνεται αμελητή επιβάλλω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε και επί της αρχής, γιατί πιστεύω εδώ καταβάλλεται συστηματικά η προσπάθεια να υπερκεράζονται κόκκινες ε, γραμμές ε, για να γίνει αποδεκτός ο ρατσισμός. Αλλά αυτό με μένα δεν θα το περάσετε. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι με βάση το άρθρο 165 του κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 11 αμελητή αποκλείεται από τις συνεδρίες και την αίθουσα ο κύριος Συναντινός. Που ακούτε κι εσείς παιδιά, τα έχω κάνει πάνω μου, ε. σας παρακαλώ. Ich fordere Sie auf, Herr Σας καλώ κύριε Συναντινέ να εγκαταλείψετε την αίθουσα και θα εισακουστείτε στο πλαίσιο της πεπατημένης. Ε, όταν λαμβάνονται αμελητή μέτρα δεν ακολουθεί συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Παρακαλώ κύριε Συναδινέ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Λυπάμαι, δεν εγκρίνω το διαδικαστικό. Κύριε Συναδινέ, παρακαλώ να φύγετε. Okay. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σας καλώ πάρα πολύ πολύ σας παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Που σημαίνει, παρακαλώ τους ε, βοηθούς ε, να απομακρύνουν τον κύριο Συναντινό από την αίθουσα. κλητήρες παρακαλώ να απομακρύνουν τον κύριο Συναντινό από την αίθουσα. Σας παρακαλώ, ε, εγκαταλείψετε την αίθουσα. Αν θέλετε να συνοδεύσετε τον κύριο Συναδίνο, εσείς, η συναδελφός του, δεν μπορώ να σας ε, εμποδίσω. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτή την απόφαση, δεν επιτρέπω διαδικαστικό. Ούτε καν να το προσπαθήσετε. Κοιτάξτε, ο κύριος Συναντινός θα εισακουστεί διακόπτει ο πρόεδρος. Κύριε Γκόλνης, εάν δεν ηρεμήστε θα σας χορηγήσουμε ηρεμιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας ε, ενημερώσω για την εξέλιξη της διαδικασίας Πρόεδρος και πάλι εφαρμόζουμε τον κανονισμό θα σας ενημερώσω για την συνέχεια της διαδικασίας. Κυρίες και κύριοι, άρχεται η ψηφοφορία. Κυρίες ε, και κύριοι, ε, πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία θα κάνω δύο ανακοινώσεις. Πρώτον, η κυρία Ελένη Θεοχάρους ε, εγκατέλειψε την πολιτική ομάδα του ΕΛΚ και από την Δευτέρα Τρίτου προσεχώρησε στην πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών